Καλημέρα συνάδελφοι. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωεκλογές. Το 2014 θα ήθελα να επενθυμίσω στους βουλευτές ότι για αυτή τη συζήτηση δεν προβλέπεται η διαδικασία του Catch the Eye. Δίνω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο Σεμέτ.